Λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσης διάταξης για τη δήλωση της Αντιπροέδρου της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΙΕΑΠ, ε, σχετικά με την κατάσταση στην Ιγυρία. Από πλευρά της ΙΕΑΠ θα ακούσουμε πάλι τον ε, Δανό Υπουργό. Ευχαριστώ και πάλι. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την κατάσταση στην Ιγυρία της ε, υπάτης εκπροσώπου αντιπροέδρου. Είναι με μεγάλη χαρά που συζητάω το θέμα αυτό. Η Νιγηρία είναι σε, μια, σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η πολιτική μεταρρυθμίσεων του Προέδρου Τζόναθαν μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της Νιγηρίας. Η δημοκρατία είναι σε φάση κατοχήρωσης και η οικονομία της αναπτύσσεται ταχαίως. Η Νιγηρία έχει τη δυνατότητα να γίνει η μεγαλύτερη οικονομία της υποσαχαρίου Αφρικής μέσα σε μερικά χρόνια. Παίζει κύριο ρόλο στην Αφρικανική Ήπειρο. Ήταν μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας πέρυσι και φέτος είναι μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο πρώην πρόεδρος ε, ο Μπαζάντζο ήταν πρόσφατα επικεφαλής της ε, οικονομικής κοινότητας των ε, δυτικοαφρικανικών κρατών και της ε, αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στον Τακάρ για να παρατηρεί τις εκλογές και να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για την Ιγυρία τους περασμένους μήνες. Το λέω αυτό με ιδιαίτερη χαρά γιατί είχα την ευχαρίστηση να εκπροσωπήσω την ΙΕΑΠ Άστον σε πρόσφατη συνάντηση υπουργική με την Ιγυρία στην Αμπούτζα στις 8 Φεβρουαρίου. Ήταν μια αξιοσημείωτη ευκαιρία και πολύ θετική. Η Νιγηρία αντιμετωπίζει ακόμη ζωτικές προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει κατηγορηματικά τις πρόσφατες επιθέσεις που διεξήγε το Μπόκο Χάραμ με την ε, απαράδεκτη απώλεια ανθρωπίνων ζώων. Οι βομβιστικές επιθέσεις κατά εκκλησιών τα Χριστούγεννα και οι πρόσφατες ε, επιθέσεις αυτοκτονίας σε μια εκκλησία στο Τζος στις 26 Φεβρουαρίου και επίσης στις 11 Μαρτίου είναι αποτρόπες. Όπως είναι και όλες οι άλλες επιθέσεις, όπως αυτή που έλαβε χώρα στο Κάνο πρόσφατα. Όλε αυτέ οι επιθέσει πρέπει να καταδικαστούν. Δυστυχώ, ο αριθμό των επιθέσεων και των ανθρωπίνων θυμάτων αυξάνεται καθημερινά. Υπάρχει μια απαράδεκτη κλιμάκωση τη βία. Η, η, η ΕΑΠ Άστον έχει εκφράσει επανειλημμένα την αλληλεγγύη τη, τη συμπαράστασή τη ε, προ τα θύματα, του τραυματίε και τι οικογένειε του. Επίση θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία να εκφράσω τη βαθιά θλίψη μας για την ε, απώλεια της ζωής των δύο Ευρωπαίων ομήρων στην Ιγυρία στις 8 Μαρτίου. Καταδικάζουμε με τους πιο κατηγορηματικούς όρους τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, όπως για παράδειγμα την ομήρια. Και από καρδιάς ε, συλληπιτήρια στις οικογένειές τους ε, για την αναντικατάστατη απώλεια που αντιμετωπίζουν. Ελπίζουμε να βρουν τη δύναμη να ξεπεράσουν τον πόνο τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τι ε, νιγηρενέ αρχέ στην καταπολέμηση τη τρομοκρατία, στην προστασία όλων των πολιτών, ιδιαίτερα των πιο ευαλώτων πολιτών και τη διατήρηση του δικαιώματο στη ζωή και του κράτου δικαίου. Οι θεμελιώδει αιτίε του Μπόκο Χάραμ είναι πολλέ. Αλλά δεν είναι σύμπτωση που έχει ισχυρότερη παρουσία στο βορρά τη χώρα, όπου έχουμε μερικού από του χειρότερου κοινωνικο-οικονομικού δείκτε στην Αφρική η βόρεια ανατολικη περιοχή της ε, Νιγηρία είναι μία από τις καταστάσεις ε, πήγουσα ανάγκη τη ξεχασμένη στον πλανήτη. Τα παράπονα των πολιτών σε αυτή την περιοχή πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να τον πιο σύντομα και εμεί ω εταίροι και φίλοι υποσχεθήκαμε στην κυβέρνηση ότι θα το κάνουμε. Τον Μποκοχάραμ επίση, επιτίθεται κατά του μη θρησκευτικού δημοκρατικού κράτου επιτίθεται κατά και των μουσουλμάνων και των χριστιανών. Η Νιγηρία παραμένει ένα μη θεοκρατικό κράτο με θρησκευτική ελευθερία που είναι σαφώ διατυπωμένη στο Σύνταγμα. Όμω, τον Μπόκο Χάραμ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τι εθνοτικο θρησκευτικέ διαφορέ που πάντα θα υπάρχουν σε μια χώρα τόσο μεγάλη με τόση ποικιλότητα όπως η Νιγηρία. τα, περί, τα περίπλοκα προβλήματα της Νιγηρίας βέβαια έχουν και θρησκευτική διάσταση αλλά δεν είναι μόνο θέμα θρησκείας ούτε ευθύνη της θρησκείας. Έχουμε έναν ε, εδρεωμένο, τακτικό διάλογο για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ιγυρία, όπου συμπεριλαμβάνουμε όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα της ελευθερίας ε, θρησκείας και συνείδησης. Η πιο πρόσφατη τέτοια συζήτηση έγινε τον Φεβρουάριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να υποστηρίξει την κυβέρνηση και το λαό της Νιγηρίας για να μην γίνεται κατάχρηση της θρησκείας για να νομοποιήσει τη βία που έχει πολιτική ή εγκληματική προέλευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ενεργή στο θέμα της ελευθερίας συνείδησης και θρησκείας, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια, σε πολλές χώρες, όχι μόνο στην Ιγυρία. Γιατί σε πολλές χώρες έχουμε διαπιστώσει μία αύξηση πράξεων θρησκευτικού μίσους και βίας. Έχουμε χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητε μας σε διμερή και πολυμερή πλαίσια στη Νέα Υόρκη και στη Γενέβη για να είμαστε πρόμαχοι στην καταπολέμηση της θρησκευτική μυσαλλοδοξία. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Όλες οι αντιπροσωπείες τη ευρωπαϊκή Ένωση παρακλήθηκαν να παρακολουθούν στενά την ε, κατάσταση στη χώρα όπου εκπροσωπούν την Ένωση και να μας κάνουν ε, εκθέσεις και να αναλαμβάνουν δράσεις. Όπως είπε, και το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών το Φεβράριο του 2011, η συνολική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό πρέπει να παρακολουθείτε από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών τους επόμενους μήνες. Ευτυχώς υπάρχουν μερικά θετικά στοιχεία. Οι Νιγηριανοί αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να βελτιώσουν την κατάσταση. Έχουμε για παράδειγμα την Ένωση των ε, Μουσουλμάνων Φοιτητών που στο Facebook καταγγέλουν τις λανθασμένες θέσεις του Μπόκο Χάραμ. Σημαντικοί ηγέτες ε, του Ισλάμ στην Ιγυρία έχουν απορρίψει τον Μπόκο Χάραμ. Λένε ότι είναι εγκληματικοί, φανατικοί που παρερμηνεύουν τη θρησκεία. Οι καθολικοί επίσκοποι επίσης έχουν λάβει θέση και επίσης η κρίση έχει αποδείξει ότι οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι στην Ιγυρία μπορούν να βοηθήσουν ένα τον άλλον και να προστατεύσουν ένα τον άλλον. Η κυβέρνηση επίσης έχει κάνει πρόοδο στην προσπάθεια εφαρμογή μιας σφαιρικής αντιτρομοκρατική στρατηγικής και διάφοροι ηγέτε του Μπόκο Χάραμ έχουν συλληφθεί. Κατά τη συνάντησή μου με την Ιγερήνη κυβέρνηση το Φεβρουάριο, του ενενθάρρυνα να βαδίσουν περισσότερο σε αυτήν την ολιστική αντιτρομοκρατική στρατηγική. Η Νιγηρία έχει μεγάλη επιρροή στον ευρύτερο κόσμο. Παίζει ένα μεγάλο σταθεροποιητικό ρόλο στην Αφρική ο τέταρτος ε, εξαγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Νιγηρία ε, δίνει ειρηνευτικές δυνάμεις στην Αφρική και είναι δυνατή η φωνή της ε, για υποστήριξη των δημοκρατιών στην περιοχή και τη ελευθερία. Οι θέσει τη Νιγηρία στι πρόσφατε κρίσει στην ακτή Λεφαντοστού και στη Λιβύη είναι σαφεί. Δηλαδή είναι ένα ισχυρό και ανοιχτό εταίρο μα στην Αφρική που από πολλές απόψεις συμμερίζεται τις απόψεις και αξίες μας. Η Υπουργική Συνάντηση είχε πολλά θετικά αποτελέσματα που θα τα προωθήσουμε περαιτέρω. Ένα είναι η συνάντηση, να, η, συγγνώμη, η απόφαση να υπάρξει τοπικός διάλογος για την ειρήνη, την ασφάλεια και την σταθερότητα και επίσης ενδιαφέρον είναι και το ενδιαφέρον της Νιγηρίας για την κλιματική αλλαγή και το Ρίο Συνήκωση. Επίσης ε, με χαράκου από τους ηγέτες στην Νιγηρία τις απόψεις του για την οικονομική ανάπτυξη. Διαφοροποιούν για να μειώσουν την εξάρτησή του από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, επενδύουν στην, ε, στις υποδομές και τη γεωργία, επικεντρώνονται στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους και για τον αυξανόμενο πληθυσμό τους 160 εκατομμυρίων ατόμων. Άκουσα πολλές φορές ότι η Νιγηρία θέλει να ενθαρρύνει επενδύσεις από την Ευρώπη και τη συμμετοχή στην ισχυρή ανάπτυξή της από την άλλη μεριά. Η Νιγηρία αντιμετωπίζει σοβαρέ προκλήσει, μεταξύ των οποίων ε, η πολύ διαδεδομένη ανέχεια. Χρειάζεται καλύτερη διακυβέρνηση, η διατήρηση τη εθνοτική αρμονία, η καταπολέμηση τη διαφθοράς και του, κρίματο είναι, του εγκλήματος συγγνώμη, είναι επίσης ε, σημαντικά καθήκοντα. Βεβαίω, το καθεστώ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ιγυρία έχει βελτιωθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχουν ακόμη τομεί όπου χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Η κατάσταση ασφαλεία στο Δέλτα του Νίγηρα, παρά το ότι έχει βελτιωθεί, παραμένει εύθραυστη. Η περιοχή είναι ζωτική σημασία για την εθνική οικονομία λόγω τη ε, παραγωγή πετρελαίου, άρα η ειρηνική ανάπτυξή τη είναι ζωτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή εφαρμόζει ένα πρόγραμμα 200 εκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσει την ανάπτυξη της περιοχής. Οι πέτρες τα τούβλα και οι λέξεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να χωρίσουν τα άτομα, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να ε, δημιουργηθούν γέφυρες. Είμαι σίγουρος ότι χάρη στις επαφές σας με τους Νιγηριανούς θα υποστηρίξετε και θα διευκολύνετε τη δημιουργία αυτών των απόλυτα ζωτικών γεφυρών που χρειαζόμαστε με την Νιγηρία και προσβλέπω στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου που θα εγκριθεί αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει από πλευράς ε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο Μάριο Μάρου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την ε, ε, μεγάλη ε, παρέμβαση με την οποία ξεκινήσατε έτσι ώστε η λεπτομερία να αναφερθείτε στην σημερινή κατάσταση στην Ιγυρία. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι δεν αναφερόμαστε μονάχα σε δύο γενικά, γενικούς ομήρους. Είναι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι, ο Μακμάρα ε, και ο Φρεντερίκο. A quella latitudine ε, και ο Φρεντερίκο Μαλινάρο. Είναι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εκεί και νομίζω ότι όπως ε, και οι Νιγηριανοί πολίτες οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι τελικά όμοιροι μιας εσφαλμένης στρατηγικής, αυτής της στρατηγικής ε, που κραδένοντας το όνομα του Θεού προσπαθεί να γονατίσει όλες τις προσπάθειες που η Νιγηρία, το κράτος, η διεθνής κοινότητα. Ε, η κοινωνία των πολιτών προσπαθεί ε, να ε, φέρει την χώρα αυτή σε ένα ηγετικό ρόλο στα πλαίσια της Αφρικής. Κύριε Υπουργέ, εγώ λέω ότι το πρόβλημα της Νιγηρίας δεν είναι οι εντάσεις, οι εθνοτικές και οι θρησκευτικές. Είναι αυτά που κρύβονται πίσω, αυτά τα παιχνίδια και οι στρατηγικές εξουσίες, που έχουν χαρακτηρίσει τους τελευταίους μήνες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό και αρνητικό τρόπο. Πρέπει να έχουμε σαφήνεια κρίσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αποτρέψουμε τον κίνδυνο της, ε, ε, ε, του εμφύλιου πολέμου. Η στρατηγική αυτών των ακραίων των ε, προσπαθούν, ε, είναι ε, ακριβώς να προσπαθούν να προχωρήσουν μέσα από τον διαστρεβλωτικό καθρέφτη της θρησκείας έτσι ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις μεγάλες, τους μεγάλους φυσικούς πόρους και αυτή τη στιγμή τελικά εκμεταλλεύονται την αδυναμία της χώρας. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ να προχωρήσετε με τις συμφωνίες τις οποίες αναφέρατε και σε αυτό θα έχετε τη στήριξη όλων μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η Βερονίκ Ντεκάιζερ από πλευρά Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι αλήθεια κύριε Υπουργέ ότι είναι δύσκολο για την Ιγυρία να φανταστεί κανείς ένα τόσο εκρηκτικό μείγμα εντάσεων. Γιατί έχουμε αφενός ε, μια εξαθλίωση και φτώχεια στο βορρά κυρίως και τεράστιο πετρελαϊκό πλούτο που τον εκμεταλλεύονται οι πολυεθνικές που ε, μολύνουν και τα ύδατα του Νίγηρα. Έχουμε και ε, συγκρούσεις θρησκευτικού χαρακτήρα μεταξύ ε, χριστιανών και μουσουλμάνων. Είχαμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις ε, του Ισμπόκο Χαράμ και την εκτέλεση, τραγική εκτέλεση δύο μύρων. Έχουμε και πολιτική διαφθορά, έχουμε κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις, αλλά πολύ σωστά μιλήσατε για τα σπάργανα μιας δημοκρατίας και μια επιθυμία της Νιγηρίας να αναλάβει τα ενία του πεπρωμένου της. Τα παράδοξα όλης αυτής της κατάστασης είναι ότι, όπως σωστά είπατε, η Νιγηρία ε, έχει ένα σημαντικό ρόλο διεθνώς ε, και στην Αφρική, ιδιαίτερα στη Δυτική Αφρική. Συμβάλλει, όπως είπατε, στην προώθηση ε, της της δυτικοευρωπαϊκής κοινότητας κρατών. Συμμετέχει σε διάφορες διαμεσολαβητικές αποστολές στο Σουδάν, στη Ζιμπάμπουε, ε, στη Νότια Αφρική, συμμετέχει σε πολλές ειρηνευτικές αποστολές και πρόσφατα μάλιστα ανέπτυξε και μια αστυνομική γυναική δύναμη στη Λιβυρία. Βέβαια, βλέπουμε την Ιγυρία που περιγράφουμε στο ψήφισμα και την Ιγυρία που ακούμε εδώ και παρατηρούμε μερικές διαφορές. Σας ζητούμε λοιπόν να απαιτήσετε από τις πετρελαϊκές εταιρείες να επιδείξουν μια διαφάνεια, να σεβαστούν το περιβάλλον και να, αποζημιώ, να καταβάλουν αποζημιώσεις για τη ρήπαση του περιβάλλοντος. Επίσης, ζητήσαμε την κατάργηση της νομοθεσίας που θεωρεί αξιόπινη την ομοφιλοφιλία. Αυτό είναι προτεραιότητα της ομάδας. Θα πρέπει να αποφυλακιστούν οι συνδικαλιστές που κρατούνται και επίσης ε, να μεριμνήσει η Νιγηρία για μια πιο ακριβοδίκαιη κατανομή του πλούτου και να σταματήσει αυτή η θρησκευτική μυσαλλοδοξία που είναι πραγματικά το φυτόριο της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σχάκ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέρυσι πήγα στην, στην για παρατήρηση εκλογών και πραγματικά ε, καλωσόριζαν τους παρατηρητές. Ήταν υποδοχή ε, πολύ θερμή και η καταμέτρηση των ψήφων έγινε με διαφάνεια. Και μάλιστα τη νύχτα πριν το πρώτο γύρο είχαμε μια έκρηξη στην Αμπουτζά που σκότωσε 25 ανθρώπους που, ετοιμάζονταν ε, που ετοιμάζονται για τις εκλογές. Οι περισσότεροι ήταν νέοι και μάλιστα συμμετείχαν σε ένα σώμα νέων. Τα παιδιά, τα παιδιά της Νιγηρίας. Και μάλιστα η βία σκοτώνει αδιακρίτως και σε συνδυασμό με τη διαφθορά και τη φτώχεια και κάποια τα προβλήματα δεν ε, ε, λαμβάνει υπόψη με ποιο τρόπο ε, θα υλοποιήσουν το στόχο τους οι εξτρεμιστές να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα και να φέρουν αντιμέτωπους ε, τους πιστούς διαφόρων θρησκειών. Η Νιγηρία φιλοξενεί ένα πέμπτο των κατοίκων της Αφρικής και πρωτοστατεί στην Αφρική. Είναι σημαντικό κράτος. 57 εκατομμύρια άνθρωποι, το μισό του πληθυσμού και είναι κάτω από 18. Δικαιούνται λοιπόν ευκαιρίες, τους αξίζουν ευκαιρίες οι νέοι της Νιγηρίας γνωρίζουν πολύ περισσότερο για τον κόσμο από ό,τι γονείς τους μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κυρίως ε, των ηλεκτρονικών μέσων. Βέβαια δεν είναι όλοι φτωχοί και δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς φτωχός σε μια τόσο πλούσια χώρα. Ε, παρακολούθησαν τα ε, αποτελέσματα των εκλογών στα κινητά τους και ζητούν λογοδοσία από τις αρχές. Δεν θα με εκπλήσει και μια άνοιξη στην Ιγυρία κάποια στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε στους νέους εκπαιδευτικές ευκαιρίες, κάτι που είναι πρόληψη, για να αποφύγουμε τη στρατολόγησή τους από εξτρεμιστικές οργανώσεις και επίσης να εξασφαλίσουμε μια οικονομική ανεξαρτησία, γιατί η Νιγηρία είναι πλούσια και από άποψη ανθρώπινο δυναμικού και από άποψη οικονομικών πόρων. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια πιο ακριβοδίκη κατανομή του πόρου, μια πιο δίκη κατανομή, μια χρηστή διακυβέρνηση για να προληφθεί ή να αναχαιτιστεί με μόνιμο τρόπο η τρομοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Από πλευρά των Πρασίνων, η κυρία Φαρτσινκίνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάνω από 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην Ιγυρία που είναι η πρώτη τρελοπραγωγός χώρα της Αφρικής και όσο πάει άσχημα η Νιγηρία τόσο αποσταθεροποιείται ολόκληρη η Αφρική. Βεβαίως η χώρα θα μπορούσε να ζει μόνο από τα έσοδα του πετρελαίου. Παρ' όλα αυτά πάνω από το 50% του πληθυσμού ζούσε, ζει σε συνθήκες ε, ε, μεγάλης ένδυας. Τα πετροδολάρια τελικά βρίσκονται μονάχα στις τσέπες ε, ορισμένων. Ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, έχουμε παραδείγματα στην Αφρική πολλά. Ε, φαίνεται ότι στην Αφρική το πετρέλαιο που θα έπρεπε να είναι ευλογία ε, γίνεται τελικά τιμωρία και πληγή ε, εμείς χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες της κυβέρνησης αλλά φαίνεται ότι υπάρχει πάντα ένα όριο το οποίο χωρίζει τους καλούς από τους κακούς αυτούς που έχουν την καλή θρησκεία από αυτούς που έχουν την κακή θρησκεία. Στην ε, ε, Νιγηρία ε, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι σκοτώνονται στο όνομα του Θεού αλλά πρέπει να ψάξουμε λίγο για να βρούμε πού ακριβώς ευθύνεται, ποιος ακριβώς ευθύνεται και ποια είναι ακριβώς η αιτία που κρύβεται πίσω από αυτή την, από αυτόν τον πόλεμο, από αυτή τη μάχη. Ε, πρέπει να απαιτήσουμε διαφάνεια ε, έτσι ώστε και το πετρέλαιο και όλα τα άλλα ε, εξορίξιμα προϊόντα να, και η διακίνησή τους να γίνεται γνωστή. όσο βελτιώνεται η κατάσταση όσον αφορά τη διαφάνεια αυτή, τόσο περισσότερο θα βελτιώνεται και η κατάσταση για τους πολίτες της Διγυρίας. Υπάρχουν πολλές Ολλανδικές εταιρείε οι οποίες παίζουν ρόλο στην ε, Νιγηρία και οι οποίες προσπαθούν να δυναμητήσουν ε, την, ε, τον κανονισμό για την διαφάνεια. Δεν θα κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Ο κύριος Τάνοκ. Τελευταία φορά μίλησα το 2010 στην Νιγηρία μετά από τη σφαγή στο Τζοζ. Και τώρα έχουμε διάφορες άλλες θηριωδίες από τον Μποκο Χαράμ και ομήρους, απαγωγές. Δυστυχώ η Νιγηρία είναι χρονικά ασταθή. Βεβαίω είναι χώρα με πολύ πληθυσμό και πολύ πετρέλαιο. Θα έπρεπε να έχει μόνιμη θέση στο Συμβούλιο ασφαλεία. Αλλά τώρα φοβόμαστε ότι μπορεί να υπάρξει εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των ε, χριστιανών και των μουσουλμάνων. Υπάρχουν εθνοτικά, πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα και εντάσει. Η κεντρική κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά αλλά δυστυχώς υπάρχει ε, πολύ εκτεταμένη διαφθορά. Επίσης υπάρχει ε, αποσχιστική ε, εξέγερση στο Νότο, στο Δέλτα του Νίγηρα. Η επιβολή του, της Σαρία σε 12 ε, ομόσπονδα κράτη στο Βορρά δημιουργεί φόβο στους χριστιανούς στο Βορρά και ίσως η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ως ενιαίο κράτος Νιγηρίας να είναι κινδύνο. Οι τελευταίες ενέργειες των ε, Βρετανών ε, κομμάντων για να απελευθερώσουν τους δύο ομήρους κατέληξαν στον τραγικό θάνατο και των δύο. Και από πλευρά της ομάδας μου απευθύνω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Τον Μπόκο Χαράμ και όλοι οι υπεύθυνοι θα πρέπει να τιμωρηθούν για την δολοφονία αυτών των δύο πολιτών της Ένωσης. Ο πρόεδρος Goodluck Τζόναθαν προσπαθεί να φέρει ασφάλεια και να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να σταματήσει τις ε, επιδοτήσεις. Να υπάρξει δηλαδή ε, ελεύθερη οικονομία στην μεγάλη νιγηριανή οικονομία. Θα πρέπει να τον υποστηρίξουμε όσο μπορούμε και οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση της βίας θα έχει τρομερές επιπτώσεις στη Δυτική Αφρική, θα δημιουργήσει τεράστιες ροές προσφύγων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη χώρα μου, το Ρωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Προβέρα, δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είδαμε, εξακολουθούν να υπάρχουν διώξεις και δολοφονίες χριστιανών. Η ένοπλη ομάδα του Μπόκο Αχαράμα που θέλει να εξισλαμίσει την χώρα έχει σκοτώσει 1.200 χριστιανούς τα τελευταία δύο χρόνια και έχει αναγκάσει 35.000 ε, χριστιανούς να εκτοπιστούν. Αλλά και σε άλλες ε, χώρες αραβικές όπως ε, η Αίγυπτος και το Ιράκ είναι χιλιάδες οι χριστιανοί οι οποίοι διώκονται ε, και εκτοπίζονται. Ε, αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα είδος θρησκευτικού ρατσισμού κατά των χριστιανών που με υποταγή και μυρολατρία φαίνεται να τον αποδέχονται όλοι. Σε αυτή την κατάσταση τα διεθνή θεσμικά όργανα συμπεριλαμβανομένες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και οι πολιτικές και θρησκευτικέ προσωπικότητες οι οποίες μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο θα πρέπει να υψώσουν τη φωνή τους έτσι ώστε οι κυβερνήσεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους και ε, θα ήθελα να πω εδώ ότι και οι λεγόμενοι μετριοπαθείς Ισλαμιστές ε, οι οποίοι δεν δέχονται τον εξτρεμισμό θα πρέπει να κατεβούν πραγματικά στην αρένα για να υψώσουν τη φωνή τους, να την ενώσουν μαζί με τους άλλους χριστιανούς. Δεν είναι δυνατόν επίσης να δεχτούμε τόσες, τόσα εκατομμύρια άνθρωποι να ζουν σε συνθήκες έσχατης φτώχειας σε μια τόσο μεγάλη, σε μια τόσο πλούσια χώρα. Όπως είπε και η συνάδελφος Αργεντίνη βεβαίως, ε, υφίσταται το πρόβλημα της μεγάλης διαφθοράς που έχει διαβρώσει όλες τις δομές της χώρας. Ε, δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά, δεν υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος, δεν υπάρχει ε, ελευθερία για το εμπόριο, δεν, υπάρχει, ε, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας για τους νέους. Στην ουσία η χώρα αυτή χρειάζεται μία σωστή και ειλικρινή και καλά προετοιμασμένη πολιτική τάξη η οποία να δημιουργήσει μια πραγματικά σύγχρονη χώρα, γιατί έτσι όπως είναι η χώρα δεν είναι ούτε σύγχρονη ούτε δημοκρατική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Εύαλτ Στάτλα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ. Ίσως να υπάρχουν ε, συγκεκριμένες συνθήκες, ε, ε, συνθήκες για την τρομοκρατία στην Νιγηρία. Υπάρχει Σαρία, υπάρχουν χιλιάδες νεκρών. Τα ξέρουμε όλα αυτά, εδώ και χρόνια δεν γίνεται τίποτα. Αλλά αυτό θα ήθελα να συμφωνήσω με τον Σνάλφο Προβέρα. Σε πολλές μουσουλμανικές χώρες, σε αυτές που είναι μάλιστα και σε άνοιξη από ό,τι λέγεται, έχουμε τρομερές διώξεις των χριστιανών. Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, στα Εμμυράτα, Πακιστάν, Συρία, στο Σουδάν. Αξιοσημείωτο. Όλο και περισσότεροι χριστιανοί υφίστανται διώξει και δεν ε, μπορούν να βρουν καμία λύση. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τολμήσει μια νέα επιθετική και αμυντική στρατηγική για να επηρεάσουμε την πολιτική στις χώρες αυτές. Δεν αρκεί να αποφασίζουμε ψηφίσματα. Βεβαίως, σωστά είναι όλα αυτά, συμφωνούμε. Αλλά δεν γίνεται και τίποτα. Το χαρτί δεν αλλάζει την κατάσταση. Η κατάσταση των χριστιανών σε αυτές τις χώρες είναι πολύ χειρότερη χρειάζονται επιγόντω τη βοήθειά μα οι χριστιανοί στι χώρε αυτέ και δεν είναι θέμα θρησκευτικών διαμαχών. Η Ευρώπη πρέπει να εκφραστεί υπέρ τη ελευθερία συνείδησης και τη θρησκευτική ελευθερία. Χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική, νέα προσέγγιση. Πώ θα μπορέσουμε δηλαδή να βοηθήσουμε του ανθρώπου αυτού, ασκώντα περισσότερη πίεση στι κυβερνήσει, ούτω ώστε να σταθούν στο πλάι των πολιτών του αυτών. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Τώρα επειδή πρέπει να φύγει δυστυχώς νωρίτερα, θα λάβει το λόγο ο κύριος Ζένταλ, εκπρόσωπος της ΙΕΑΠ, και μετά θα πάρει το λόγο για να κλείσει συζήτηση ο Επίτροπος κύριος Πίμπαλ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη για αυτή την άκομψη κατάσταση, αλλά ε, ε έχω και υποχρεώσεις κυβέρνηση της χώρας, επομένως πρέπει να φύγω. Ε, σχετικά με την συζήτηση αυτή πρέπει να ομολογήσω ότι υπήρξε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, σας μίλησα προηγουμένως και για την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Ιγυρία και Προσπάθησα να σας μεταφέρω τις εντυπώσεις μου. Βεβαίως ε, θα είναι εδώ ο Επίτροπος ο οποίος θα απαντήσει στις περαιτέρω ερωτήσεις σας. Πάντως θα ήθελα να σας πω ότι εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος ε, να έχει κάποιο όφελος από αυτήν την θρησκευτική διαμάχη είναι μόνο η οργάνωση Μπόκο Χαράμ. Δεν πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι τους. Ε, δεν πρέπει να τους αφήσουμε ε, να κυριαρχήσουν σε μια χώρα ε, που έχει διαφοροποιημένη πολιτιστική κατάσταση όπου υπάρχουν πολλές διαφορετικές θρησκείες ε, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να παίξουμε το θρησκευτικό παιχνίδι της οργάνωσης Μποκοχαράμ. Ε, τούτου λεχθέντος πάντως θα πρέπει οι, όλες ε, οι θρησκείες να προστατεύονται. Θα πρέπει οι πιστοί όλων των θρησκειών να μπορούν να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα με ελευθερία. Αυτή τι ε, που μας απασχολούν περισσότερο είναι οι μουσουλμάνοι του Βορρά, ε, γιατί εκεί φαίνεται να γίνονται ε, οι περισσότερες θρησκευτικές ζυμώσεις. Ε, τα πρόσφατα ε, γεγονότα ε, οπωσδήποτε μας τρόμαξαν όλους και εμείς εκφράσαμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια για τις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους. Καταδικάζουμε τέτοιες κινήσεις Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες οι οποίες δολοφονούν ε, ανθρώπους και δεν μας ενδιαφέρει ε, ε, πίσω από ποια ιδεολογία διαπράττονται τα εγκλήματα αυτά. Εξακολουθούν να είναι εγκλήματα. Δεν μπορεί κανείς να αφαιρέσει τη ζωή κάποιου άλλου για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να συρθούν ενώπιον των δικαστηρίων και κυρίως να μην παρουσιάζονται σαν μάρτυρες. Είναι εγκληματίες, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφαιρέσει αφαιρέσει τη ζωή άλλων ανθρώπων. Ε, να δώσω και κάποιες επιπλέον ε, πληροφορίες. Ελπίζω ότι θα έχω την ε, δυνατότητα να σας δώσω σύντομα. Σύντομα δηλαδή θα συναντηθώ με τον πρόεδρο της Νιγηρίας και ελπίζω ότι από την επίσκεψη και τη συνάντηση αυτή θα επιστρέψω με περισσότερες πληροφορίες και ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε μια Αφρικανική χώρα η οποία έχει υψηλό ηθικό και η οποία θέλει να προχωρήσει Έχουμε επίσης, και δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό, να κάνουμε με μια χώρα ε, ε, με πολύ νεανικό πληθυσμό που ε, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, κυρίως δε το πρόβλημα της τρομοκρατίας στο Βορρά. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει στεναρά την κατάσταση αυτή κυρίως για να βοηθήσει τους πιο φτωχούς πολίτες της. Η κατάσταση πάντως είναι ιδιάζουσα. Ε, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πιστεύουμε ότι η Νιγηρία μπορεί και πρέπει να παίξει σταθεροποιητικό ρόλο στην ε, Αφρική γενικότερα και στη Δυτική Αφρική ειδικότερα. Δεν πρόκειται για μια φτωχή χώρα και επομένως απλά θα πρέπει ε, να καταπολεμήσει την διαφθορά έτσι ώστε όλοι να μπορούν να έχουν μερίδιο στον πλούτο. Είναι βέβαια επικίνδυνο έργο αυτή η καταπολέμηση της διαφθοράς. Ε, η κυβέρνηση είναι νέα και πρέπει να της δώσουμε και λίγο χρόνο. Ε, πάντως πρόκειται για ένα θέμα το οποίο εξακολουθεί να μας απασχολεί ε, και θα τελειώσω λέγοντας ότι η χώρα αυτή θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο δημογραφικό βάρος τα επόμενα χρόνια. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν να μας απασχολήσει με μεγάλη σοβαρότητα. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και τώρα Περνάμε στους επόμενους ομιλητές. Η κυρία Όμεν Ράιτεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ο αριθμός των τρομοκρατικών επιθέσεων, όπως μας ανέφεραν και οι συνάδελφοι, ήταν μεγάλος και οι τρομοκρατικές αυτές επιθέσεις ε, έγιναν κυρίως από μέλη της ε, οργάνωσης Boko Haram, ο φόρος σε ανθρώπινες ζωές ήταν πολύ βαρύς. Και ο τρόπος αυτός χρησιμοποιήθηκε από την ένοπλη οργάνωση Μπόκο Αράμ για να αποσταθεροποιήσει τη χώρα. Η κοινωνική αδικία, η εξαθλίωση, η φτώχεια, η διαφθορά, η... το υψηλό ποσοστό ανεργίας και η έλλειψη προοπτικής για τους νέους ε, δημιουργούν ένα πρόσφορο έδαφος για τον εξτρεμισμό. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο οφείλει να καταδικάσει δρυμύτατα και απερίφραστα τη βία, αλλά να κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει τη χώρα αυτή στις προσπάθειές της. Και είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο αυτό είναι η διεθνής κοινότητα να επικεντρωθεί στα αίτια του κακού, στα, στις ρίζες αυτής της κατάστασης. Γιατί μια τόσο πλούσια χώρα όπως είναι η Γυρία να μην μπορεί να ε, μοιράσει αυτό το πλούτο στους πολίτες της. Θα πρέπει να ενισχύσουμε και τη διαπεριφερειακή συνεργασία. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς στη διαδικασία αυτή. Κατάλαβα ότι ο, την περασμένη εβδομάδα ο Ολλανδός Υπουργό Εξωτερικών ζήτησε να τεθεί η οργάνωση Boko Haram στον κατάλογο με τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Διαρωτώ με αν ε, συνέβη τελικά κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Κορτές Λάστρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να καταδικάσω καταρχήν τη βία των τελευταίων μηνών στην Ιγυρία. Η Ιγυρία είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της ε, Αφρικής και με τις καλύτερες ε, οικονομικές προοπτικές ε, και για αλλοδαπές επενδύσεις. Είναι χώρα που εξάγει πετρέλαιο και έχει τεράστιους πόρους και πλούτο που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει για να καταπολεμήσει την ανισότητα και τη φτώχεια που μαστίζει τη χώρα. Κύριε Επίτροπε, σε πολλές περιπτώσεις ε, τα μέλη της Επιτροπής ανάπτυξη τάχθηκαν υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπέρ τη Δημοκρατία ε, και είπαμε ότι αυτά συνδυάζονται με την ε, δημοκρατία και την ανάπτυξη. Οι ρίζε τη σύγκρουση στην Ιγυρία βρίσκονται στην εξαθλίωση και τη φτώχεια στην οποία είναι βυθισμένη ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Δυστυχώ ο πλούτο τη χώρα δεν είναι σωστά κατανεμημένο ε, στα πιο φτωχά τμήματα του πληθυσμού. Γι' αυτό και εκατομμύρια Νιγηριανοί είναι ευάλωτοι και δεν έχουν πρόσβαση στι στοιχειώδει ε, υπηρεσίε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη αναπτυξιακή τη πολιτική και πολιτική συνεργασία μπορεί να κάνει διαφορά, τη διαφορά στη χώρα. Θα πρέπει να έχουμε μια κοινή στρατηγική καταπολέμηση τη φτώχεια και καλύτερη πρόσβαση στις στοιχειώδει υπηρεσίες όπως είναι η υγεία και η εκπαίδευση για τα πιο ευάλωτα άτομα. Η προστιθέμενη αξία τη Ευρωπαϊκής Ένωση, για τη χώρα αυτή θα είναι να μειώσει τις ανισότητες και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας να φέρει όλο και περισσότερους ε, ανθρώπους από την ε, εξαθλίωση και τη φτώχεια σε ένα πιο υψηλό βιωτικό επίπεδο. Δεν αρκεί όμω μια τέτοια πολιτική. Θα πρέπει να είναι συνεπή μα η αναπτυξιακή πολιτική με τι υπόλοιπε μα πολιτικέ απέναντι στην Ιγυρία. Πολύ σημαντική είναι επίση ε, η διαφάνεια που θα πρέπει να διέπει τι ε, εργασίε των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ιγυρία. Ελοχεύει ένα σοβαρότατο κίνδυνο στην Ιγυρία και γενικότερα στην Δυτική Αφρική και στην ε, περιοχή του Σαχέλ. Είχαμε παρατεταμένη ε, ανοβρία, μικρές ε, σοδιές, με λίγα ζώα στην κτηνοτροφία και η αύξηση των τιμών των τροφίμων δημιουργεί πολύ ζωφερέ προοπτικές για την Ένωση. Οι οργανώσεις του ΟΗΕ και οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών μας προειδοποιούν για αυτή την επικείμενη τραγωδία. Θα πρέπει να αντιδράσουμε λοιπόν εγκαίρως και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τη λιμοκτονία πριν θερήσει περισσότερες ζωές στην περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χωρίς να θέλω να πάρω βραβείο πρωτοτυπίας, πρέπει να σας πω και εγώ ότι στην Νιγηρία το έδαφος είναι πρόσφορο ε, για τέτοιου είδους ε, τρομοκρατικές ε, ενέργειες ο, οι ε, Ισλαμικοί, οι Ισλαμιστές ε, εξτρεμιστές ε, προσπαθούν να τρομοκρατήσουν εθνοτικές μειονότητες και άλλες θρησκείες. Όλα αυτά συμβαίνουν παρά το μάνα του πετρελαίου που θα έπρεπε να αλλάξει την κατάσταση. Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σταθεροποιήσουν την κατάσταση στο Δέλτα του Νίγηρα και για να βελτιώσουν την διακυβέρνηση, τα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς είναι οπωσδήποτε σωστά, αλλά βεβαίως πρώτες οι νιγηριανές αρχές είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάμπερτ, παρακαλώ. Κυρία Λάμπερτ, συγγνώμη, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρετίζω αυτή την ευκαιρία. Επιτέλου, να κάνω μια συζήτηση για την Ιγυρία. Είναι πολύ σημαντική χώρα, όπω ακούσαμε. Πολύ σημαντική στην περιοχή, αλλά και παγκοσμίω. Λυπάμαι ότι ο μόνο τρόπο που συζητάμε στη, για την Ιγυρία είναι και πάλι μέσω ψηφίσματος που ε, ενοχοποιεί τη θρησκεία. Να απαντήσω σωσμένα από όσα υπόθηκαν. Να είμαστε σαφείς. Το Μπόκο Χαράμ είναι κυρίως υπεύθυνο για τη βία, αλλά δεν σκοτώνουν μόνο χριστιανούς. Έχουν σκοτώσει και μουσουλμάνους που δεν συμφωνούν μαζί τους. Επίσης υπήρξαν ε, δολοφονίες ε, μουσουλμάνων ως αντίπεινα από τους χριστιανούς, λεγόμενους χριστιανούς. Έχουμε δει πολλούς ηγέτες και θρησκευτικούς και πολιτικούς από διάφορες ε, τοποθετήσεις και απόψεις να καταδικάζουν τη βία. Είναι σημαντικό λοιπόν να τονίσουμε αυτά που ενώνουν αυτή τη χώρα, όχι μόνο αυτά που τη διαιρούν. Βεβαίω, η διαφθορά είναι μεγάλο θέμα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Καλωσορίζω την πρόσφατη την ε, πρόσφατη δίκη του Ιμπόρη, πρώην ε, κυβερνήτη του ομόσπονδου κράτου ε, του Δέλτα του Νίγηρα, σε Βρετανικό δικαστήριο που είναι τώρα στη φυλακή. Μπορούν όμω να γίνουν περισσότερα για την καταπολέμηση τη διαφθορά. Η κυβέρνηση η, πρέπει όμω να μπορεί να παίξει το ρόλο τη. Γι' αυτό είμαστε διατεθειμένοι. Συγγνώμη, είναι διατεθειμένοι οι πολίτε τη Νιγηρία να κάθονται ώρε στον ίδιο για να μπορέσουν να ψηφίσουν. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει η Ένωση τη σχέση τη με την Ιγυρία. Το κοινοβούλιο μα πρέπει να ενισχύσει τι σχέσει του με το Ιγυριανό κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ τον κύριο Σιμάνσκι. Α, δεν τον βλέπω εδώ. Οπότε, ο επόμενος ομιλητής για 1,5 λεπτό, κύριος Μπέλντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η Ισλαμιστική και η τρομοκρατική οργάνωση Boko Haram ε, είναι μονάχα μία από τις οργανώσεις που δρούν στην ε, Νιγηρία ε, και η κατάσταση των χριστιανών ε, γίνεται όλο και πιο δύσκολη γιατί αποτελούν αντικείμενο σημαντικών διώξεων και θα πρέπει να προστατευτούν. Η βία της οργάνωσης Boko Haram είναι πάρα πολύ μεγάλη και επιτίθεται κατά όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων του Βόρειου τμήματος της ε, χώρας. Οι απώλειες είναι πολύ μεγάλες ε, και ακόμα αυτός ο κύκλος της βίας δεν έχει σταματήσει. Θα έχουμε ακόμα πολλά θύματα. Πρόκειται εδώ ε, για προστασία όλων των θρησκειών και ε, ε, βεβαίως ε, θα πρέπει αυτό να γίνεται σαφές παντού. Επίσης θα πρέπει να μελετήσουμε το κατά πόσον έχει καταφέρει να βάλει τα πλοκάμια της Ιμπόκο Χαράμ και στην κυβέρνηση της Νιγηρίας. Είναι μια ερώτηση που θέλω να απευθύνω στον Επίτροπο και θα απευθύνω και στην ίδια την κυρία Άστον όταν θα εμβαθύνει ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Το ε, ε, έχει γνώση σχετικά με αυτό το θέμα, δηλαδή κατά πόσον η Μπόκο Χαράμ έχει παρισφρήσει εις ε, την κυβέρνηση. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον η Μπόκο Χαράμ δουλεύει και μέσα από κάποιες οργανώσεις της Μεγάλης Βρετανίας. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντόντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατάγομαι από τη Βόρεια Ιρλανδία και γνωρίζω πολύ καλά το φόβο και το πόνο, την οδύνη που βιώνουν οι Γυριανοί εξαιτία τη κλιμακούμενη βία κάποιων τρομοκρατικών ομάδων που σκοτώνουν του ανθρώπου μόνο και μόνο λόγω τη θρησκεία του. Και μάλιστα οι περισσότεροι ε, Νιγηριανοί ζουν από το φόβο των τρομοκρατικών ε, ε, επιθέσεων. Μόνο το Φεβρουάριο το Τζος, στο Τζο σκοτώθηκαν τρει άνθρωποι από βομβαρδισμό μια εκκλησία. Αυτέ ήταν από τι τελευταίε βομβαρδιστικέ επιθέσει. Οι τρομοκράτε επιτίθενται σε μια εκκλησία μόνο και μόνο επειδή είναι εκκλησία και θα αποφασίσουν να επιτεθούν σε οποιαδήποτε εκκλησία. Τώρα έχουν ξεκινήσει. Φαίνεται ότι οι πολεμοχαρείς Ισλαμιστέ τη Μπόκο Χαράμ θέλουν να εξολοθρεύσουν το χριστιανικό πληθυσμό της Νιγηρίας. Βέβαια, συμφωνώ με αυτό που είπαν οι συνάδελφοι, ότι και άλλοι μη χριστιανοί έχουν υποφέρει και έχουν χάσει τη ζωή τους. Φυσικά καταδικάζω ως ηλίδιν όλες αυτές τις επιθέσεις. Το να χάνει κανείς τη ζωή του λόγω της θρησκείας είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είναι μόνο θέμα φτώχειας ή διαφθοράς. Εδώ μιλούμε για επίθεση κατά συγκεκριμένου τμήματος της κοινωνίας της Νιγηρίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Κατσμάρεκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Το 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ενέκρινε ένα ψήφισμα που στυλίτευε τις μαγικές σφαγές στα περίχωρα της Γιος ε, που διαδραματιζόταν τότε πραγματικό πογκρόμ κατά των χριστιανών. Βέβαια η κατάσταση δυστυχώ έχει επιδεινωθεί στην ε, Νιγηρία. Η ανεξιθρησκεία βέβαια τυπικά κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα, αλλά δυστυχώ ε, η κρατική εξουσία είναι ανήμπορη να αντιμετωπίσει την οργανωμένη εγκληματικότητα που δεν αποδέχεται αυτή την ελευθερία. Η οργάνωση Boko Χαράμ τρομοκρατεί του χριστιανού ε, και προσπαθεί να επιβάλλει τον Ισλαμικό νόμο σε όλα τα ομόσπονδα κρατήδια τη Νιγηρία προσφεύγει σε βομβιστικές επιθέσεις όπου έχασε τη ζωή τους 900 άτομα και μάλιστα εκτελέστηκαν και δύο όμοιροι, ένας Βρετανός και ένας Ιταλός μετά από κράτηση 10 μηνών. Πριν από δύο χρόνια είχαμε κάποιες αμφιβολίες κατά πόσο κύριο αίτιο για τα έκτροπα στην Ιγυρία, είναι η θρησκεία. Οι, ε, οι θεωρούν ότι οι αιτίε τη βία στην Αιγυρία είναι περίπλοκες, οικονομικές, κοινωνικές, εθνοτικέ και πολιτισ, πολιτιστικές. Ο λόγος πάντως για τους βιασμούς στην Ιγυρία είναι η θρησκευτική μυσαλλοδοξία. Μπόκο Χαράμ σημαίνει ε, δυτική ανατροφή είναι αμαρτία και η εντολή για πάταξη της ε, αμαρτίας έχει, έχει θρησκευτικό χαρακτήρα. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε στην Ιγυρία εκείνους που προσπαθούν ε, να, να αντιταχθούν στο θρησκευτικό φανατισμό. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κ. Ευχαριστώ πολύ. Μας απασχολεί όλους, ε, μας απασχολεί πολύ η κατάσταση στην Ιγύρια. Ε, τον ε, Φεβρουάριο ακόμα σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Είχαμε επίσης και τις εχμαλωσίες ανθρώπων, καθώς επίσης και τα τραγικά συμβάντα της, του τελευταίου Σαββατοκύριακου με την απώλεια τριών ανθρώπινων ζωών. Μας απασχολεί το θέμα αυτό, ενώ φαίνεται ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία ε, για να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να ξεκινήσει έναν ε, καλό διάλογο ανάμεσα στις κοινότητες και τις ε, θρησκείες. Ο πλούτος της Νιγηρίας θα έπρεπε να οδηγεί στην ευζοία των κατοίκων, ενώ συμβαίνει τελικά το αντίθετο. Το πετρέλαιο φέρνει τελικά μόνο προβλήματα, εχμαλωσίες, απαγωγές ξένων, περιβαλλοντική μόλυνση κτλ. Μπορούν και οι πολίτες να παίξουν ρόλο για τη σταθεροποίηση της χώρας ε, και βεβαίως δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε πλέον ε, τα ε, χρήματα, τα ωφέλη από το πετρέλαιο να βρίσκονται μόνο στις τσέπες μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών όπως ας πούμε η Shell. Θα πρέπει να είναι αρκετά δυνατές οι αρχές, να είναι αρκετά δυνατή η κυβέρνηση και να προχωρήσει σε σημαντικές αποφάσεις όσον αφορά τη φορολογία και επίσης όπως είπε και η κυρία Σαρτζεντίνη να ενεργοποιήσουμε και τις ερήτρες διαφάνειας η ελευθερία, η ηρεμία, η ενεξιθρησκεία είναι στοιχεία εξαιρετικά ε, σημαντικά τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η ύπατη εκπρόσωπος θα πρέπει να παρέμβει έτσι ώστε οι αρχές αυτές ε, να λειτουργήσουν στη χώρα και ώστε να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή να τις εφαρμόσει. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μεταξύ των διαφόρων ατυχιών της Νιγηρίας ε, καταγράφεται και η δολοφονία των Φράνκο Λαμολινάρα και, και, του ε, Είναι λυπηρό το γεγονός ε, του, του θανάτου της, αλλά ε, λυπηρός είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το πρόβλημά τους σε επίπεδο ασυνεννοησίας στο Ευρωπαϊκό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητέ κύριε Επίτροπε. Θέλω να πω στον Επίτροπο ότι οι Ευρωπαίοι, οι πολίτες θέλουν να βλέπουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουν οποτεδήποτε συμβαίνει κάτι στο εξωτερικό, όπως ας πούμε στην Ιγυρία, ε, να είναι συγκεκριμένη η αντίδραση. Ε, ε, σε αυτήν την περίπτωση Ιταλοί δεν ειδοποιήθηκαν καθόλου και συμμετείχαν μονάχα οι Βρετανοί σε μια τελικώ αποτυχημένη ε, προσπάθεια. Ζητούμε από την Ιγυρία να καταβάλει και αυτή η μεγάλη προσπάθεια, αλλά βεβαίω θα πρέπει να δούμε και τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αποτρόπη βία της ε, οργάνωσης Μποκοχάραμ ήδη περιγράφηκε από τους συναδέλφους. Ε, είναι αποτρόπη και με την εκτινοδία τους ε, μπαίνουν στις σελίδες των μέσων ενημέρωσης. Πρόκειται για άθλιες πράξεις βίας. Τον Ιούλιο του 2009 δολοφονήθηκαν πάνω από 700 άτομα. Στο Πλατιάο, το τομός κράτος, το 2010 υπήρξε βία για λόγους θρησκευτικούς με 300 θύματα και 10.000 εκτοπισμένους. Υπήρξε μια επιτροπή έρευνας της κυβέρνησης, υπήρξε μια έκθεση, αλλά ούτε το 2009, ούτε το 2010, ούτε πριν το 2008 οι, δημοσιεύτηκαν αυτές οι εκθέσεις και ούτε δόθηκαν τα ονόματα των ε, υπευθύνων. Είναι σοβαρές παραλήψεις αυτές. Θέλω να το υποστηρίξω. Γιατί το αναφέρουμε και στο ψήφισμά μας δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτέ οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατόπιν να μην υπάρχουν συνέπειε. Θέλω να το αναφέρω αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό έχει τώρα ο κύριο Τσιόμπρο. Μικρό, πείτε. Ευχαριστώ. Στα μάτια μας ε, ε, ε, διαδραματίζεται στην Ιγυρία μια τραγωδία. Άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, είναι θύματα μιας θρησκευτικής θηριωδίας. Οι μουσουλμάνοι δολοφονούν χριστιανούς μόνο και μόνο επειδή πρεσβεύουν άλλη θρησκεία με διαφορετικό τρόπο ε, αντιμετωπίζουν την παράδοση και τις αξίες τους. Είναι πραγματικά ε, τραγικό να διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια μας τέτοιες τραγωδίες. Οι συγκρούσει ε, μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων δεν είναι καινούριε. Δυστυχώ όμω η διεθνή κοινότητα δεν αντέδρασε έντονα. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτής της μυσαλλοδοξίας τα είδαμε και την περασμένη Κυριακή όταν ε, στο γιος με βοβηθιστική επίθεση της Μποκοχαράμ έξανε τη ζωή του τρεις αθώοι άνθρωποι. Θα πρέπει να καταδικάσουμε απερίφραστα το, την Ισλαμική τρομοκρατία εις βάρος των χριστιανών και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τι συγγυριανές αρχές να σταματήσουν αυτό το μακελιό και την αιματοχυσία και να επαναφέρουν τη χώρα στο σωστό δρόμο. Δυστυχώ αυτό λείπει σήμερα, μια αποφασιστική και απερίφραστη καταδίκη του Ισλαμικού εξτρεμισμού στην Ιγυρία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μίτσουλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι ενέργειες του Μπόκο Χαράμ είναι αποτρόπες, φανατικές, είναι πράξεις ε, μίσους. Πρέπει να δεσμευτούμε να τιμωρηθούν μέσω της δικαστικής οδού. Καλό την ΙΕΑΠ να υπάρξουν διακανονισμοί ούτω ώστε να καταλάβουν ότι όντως θα τιμωρηθούν. Ε, από το 2009 η ομάδα αυτή προσπαθεί να ανατρέψει την κυβέρνηση της Νιγηρίας εκατοντάδες θύματα, βομβιστικές επιθέσεις. Και τώρα έχουν διευρύνει τους στόχους τους. Όχι μόνο η αστυνομία και οι δημόσιες αρχές, μόνο απλοί χριστιανοί που πηγαίνουν στην εκκλησία. Έχουν κάψει εκκλησίες στην πόλη του Τζος, σκότωσαν εκεί 185 άτομα όπως ακούσαμε. Σε οποιαδήποτε κοινωνία αυτό είναι τελώς απαράδεκτο. Αλλά αναφέρω και το γεγονό ότι η Νιγηρία είναι ο 8ο παραγό πετρελαίου στον κόσμο. Και όμω ε, η πλειονότητα των 145 εκατομμυρίων κατοίκων, κατοίκων τη Νιγηρία ζουν κάτω από την, ε, το επίπεδο τη φτώχεια. Αυτό πρέπει να το θίξουμε. Όχι μόνο έναντι τη κυβέρνηση, αλλά και του παραγωγού, αυτού που εκμεταλλεύονται αυτό το πετρέλαιο. Πρέπει να κυνηγήσουμε αυτού που κάνουν αυτά τα εγκλήματα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να επηρεάσουμε και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το θέμα η παραγωγή πετρελαίου. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Κρέτσου. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που συμβαίνει στην Ιγυρία, η αστάθεια, ο εξτρεμισμός, η βία είναι πολύ σοβαρά και δύο πολίτες των χωρών μας ε, θανατώθηκαν. Ε, πρέπει λοιπόν να κρούσουμε έντονα τον κόδωνα κινδύνου. Δεν πρέπει να επεκταθεί αυτή η βία μεταξύ των θρησκειών στην Αφρική. Πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν τρομοκρατικές ομάδες σε αυτή την περιοχή που συντονίζουν τη δράση τους με την Αλκάιντα. Πρέπει να μας ανησυχήσει περισσότερο η Νιγηρία. Γιατί είναι η μεγαλύτερη χώρα από πλευρά πληθυσμού τη Αφρική. 160 εκατομμύρια κατοίκου. Εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι πολύ φτωχοί. Ακόμη και αν η χώρα δεν είναι καθόλου φτωχή. Η Νιγηρία είναι ο δεύτερο πετρελοεξαγωγό του κόσμου και είναι παράλληλα μία από τις πιο διεθαρμένες χώρες σύμφωνα με την ε, κατάταξη που μπορούμε να δούμε. Και επίσης ε, η ανάπτυξη των ανθρώπων είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εκλογές, να επιτηρήσουμε σε όλες τις χώρες Αφρικής, ώστε να καταργήσουμε την ε, διαφθορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτρελε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε πίτροπε. Κυρίες και κύριοι, πέρυσι κατά τη διάρκεια των εκλογών είχα την ευκαιρία να μεταβώ στην ε, Νιγηρία και να τη γνωρίσω καλύτερα. Είναι από του σημαντικού εταίρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και λυπούμε που αμέσω μετά τι εκλογέ είχαμε τρομοκρατικέ επιθέσει και γενικώ βίε εξάρσει που αποσταθεροποίησαν τη χώρα. Παρατηρούμε μία έξαρση δυστυχώ τη τρομοκρατία. Είμαι πεπισμένο ότι οι σχέσει μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών δεν είναι εσωτερικό μόνο ζήτημα τη συνηγυρία. Ξέρω ότι η πλειοψηφία και των χριστιανών και των μουσουλμάνων είναι υπέρ μιας βιώσιμης δημοκρατικής ανάπτυξης της Νιγηρίας. Τρία είναι τα πιο σημαντικά για το μέλλον της Νιγηρίας, δηλαδή η βελτίωση της διακυβέρνησης, η λήψη υπόψη των αναγκών των διαφόρων περιοχών, η συστηματική ε, αντιμετώπιση των ε, αιτίων και των πηγών των συγκρούσεων και φυσικά η αποφυγή της χρήσης βίας ή η βία επιβολή μιας πολιτικής βούλησης. Καλό θα ήταν να ενισχύσουμε την συνεργασία μας με την Ιγυρία και να αναπτύξουμε και τον, την κοινοβουλευτική διάσταση αυτής της συνεργασίας. Θα ήθελα να χαιρετήσω εδώ τον αξιοχότατο πρέσβη της Ιγυρίας, τον κύριο Μπαράια, που παρακολουθεί τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πέτερλε. κυρία Στριφλέα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπή, αγαπητοί συνάδελφοι. Το κοινοβούλιο μα πρέπει να καταδικάσει κατηγορηματικά την πρόσφατη βία στην Ιγυρία, ιδιαίτερα τι τρομοκρατικέ επιθέσει που έγιναν από το... την Ισλαμιστική σέκτα Μπόκο η απόλυτη φτώχεια, η διαφθορά, η ενδημική διαφθορά, η κακή διακυβέρνηση διαμορφώνουν ένα κατάλληλο κλίμα για αυτή την εξτρεμιστική οργάνωση μπορεί να στρατολογήσει πολύ εύκολα μεταξύ των νέων ανέργων η κυβέρνηση της Νιγηρίας πρέπει ταχύτατα να πάρει αποτελεσματικά μέτρα για να προστατεύσει τους πολίτες της, να σταματήσει αυτή η γενικευμένη διαφθορά ή ασυδοσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει την κυβέρνηση στις προσπάθειες αυτές. Πιστεύω επίσης ότι δεν πρέπει να απλοποιούμε τις συγκρούσεις, να λέμε ότι οφείλεται μόνο στη θρησκεία αυτή η βία. Πρέπει να καταλάβουμε τις εντάσεις που υπάρχουν στην Νιγηρία, που έχουν οικονομική και κοινωνική διάσταση. Η Νιγηρία είναι ο πιο μεγάλος ε, παραγωγός αργού πετρελαίου στην Αφρική, αλλά αυτός ο πλούτος δυστυχώς γίνεται αντικείμενο πολύ κακής διαχείρισης. Οι αρχές της Νιγηρίας, αλλά και οι πολυεθνικές του πετρελαίου, πρέπει σύντομα να μειώσουν, να καταργήσουν, να αντιμετωπίσουν και να εξαλείψουν την ε, μόλυνση που προκαλεί το πετρέλαιο στο περιβάλλον και που είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για τον πληθυσμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Κύριος πρέτα Κριστιαν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και πολλούς μήνες Ακούμε δυστυχώ πολύ ζωφερέ ειδήσει από την Ιγυρία που γίνονται όλο και πιο ανησυχητικέ. Οι δράσει τη τρομοκρατική οργάνωση Μπόκο Χαράμ γίνονται όλο και πιο βίες. Τον Νοέμβριο του 2011, 55 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του σε μια σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ταματούρ. Και την ημέρα των Χριστουγέννων, 44 άτομα έχασαν τη ζωή του στην τρομοκρατική επίθεση σε μια καθολική εκκλησία τη Αμπούτζα. Και μάλιστα οι τρομοκρατικές επιθέσεις ε, στο Κάνο, στα βόρεια της Νιγηρίας, ε, έφεραν το θάνατο σε 185 άτομα. Είναι από τις πιο βάρβαρες και αποτρόπες ενέργειες και πράξεις που διεκδίκησε η Μπόκο Χαράμ. Εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες μάλιστα, η Νιγηρία ε, είναι πεδίο σύγκρουση μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Η ένταση πια είναι προφανή, δεν μπορούμε να την αγνοούμε και οι συγκρούσεις αυτές απειλούν τη σταθερότητα του συνόλου της χώρας. Όλο και περισσότεροι ζητούν, αναρωτιούνται πια μήπως η Νιγηρία μπήκε σε μια πολύ ε, ε, μοιραία πορεία εξαφάνισης. Θα πρέπει να επαναφέρουμε την ανεξιθρησκεία στην, στην Ιγυρία. Επίσης θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο εδάφιο 7 του κοινού ψηφίσματος, γιατί η Μπόκο Χαράμ δεν απειλεί μόνο την Ιγυρία, αλλά και την ευρύτερη περιοχή εξαιτίας των πιθανών διασυνδέσεών της με την ΑΚΜΗ. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη διαπεραφερειακή συνεργασία και τις προσπάθειες ε, για να αποφευθεί η συνεργασία Μποκοχαράμ και ΑΚΜΗ. Ο κύριος Σόνικ. Ευχαριστώ. Η βία με θρησκευτικό και εθνοτικό υπόβαθρο ε, ε, έφερε σε, θάνατο δεκάδες, ε, εκατοντάδες ανθρώπους στην Ιγυρία την τελευταία δεκαετία και μάλιστα τον τελευταίο καιρό δυστυχώς είχαμε κλιμάκωση της θρησκευτικής βίας εξαιτία των ενεργειών τη τρομοκρατική οργάνωσης Ποκοχαράμ. Τον Ιούλιο το, το 2010 η Μπόκο Χαράμ είχε ε, 160 ε, τρομοκρατικές επιθέσεις ε, και ε, έχασαν τη ζωή τους εκεί 900 περίπου άτομα. Προσπαθεί η Μπόκο Χαράμ να εφαρμόσει τον Ισλαμικό νόμο και σε 36 ομόσπονδα κρατήδια της Νιγηρίας. Και μάλιστα απειλεί τους τους χριστιανούς με εκτοπισμό από τη χώρα. Οι χριστιανοί είναι από τις ε, πιο ε, κατατρεγμένες θρησκευτικές ομάδες της Νιγηρίας και απειλούνται με εξολόθρευση. Θα έχουμε μαζικές μεταναστεύσεις αν γενικευτεί αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς ε, επικρατεί και μια πολιτική αστάθεια στην Ιγυρία και σημαντική διαφθορά που οδηγεί σε μια πολύ άνηση κατανομή του πλούτου. Είναι από τις πιο πλούσιες χώρες η Νιγηρία με το σημαντικότερο ΑΕΠ εξαιτία του πετρελαίου, αλλά δυστυχώς ε, ένα συντριπτικό ποσοστό του πληθυσμού ε, ζει σε ε, επίπεδο εξαθλίωση με λιγότερο από 2 δολάρια την ημέρα. Φυσικά έχουμε και τον θρησκευτικό φανατισμό στο υπόβαθρο αυτό. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν το διάλογο με την κυβέρνηση της Νιγηρίας ώστε να εξασφαλίσουμε μια τάξη που θα είναι και δίκαιη στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Βένσον, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Δανός Υπουργό ε, στις σύντομες ε, καταληκτικές παρατηρήσεις του για την Ιγυρία αναφέρθηκε στους πολιτικούς ηγέτες και είπε ότι είναι καλή. Ίσως και να είναι, αλλά είναι ντροπή μια τόσο πλούσια χώρα με τόσο πετρέλαιο να είναι τόσο διεφθαρμένη και η φτώχεια να είναι τόσο διαδεδομένη και να θίγει τόσο μεγάλο τμήμα του πληθυσμού σε μια τόσο πλούσια χώρα με τέτοιους ε, φυσικούς πόρους. Μιλήσαμε για τι εντάσεις μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Κανεί δεν μπορεί να ξεφύγει από τα αποτελέσματα αυτών των εντάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δίνει βοήθεια μέσω πενταετών προγραμμάτων, ε, διάφορα εκατομμύρια ευρώ. Θα θέλαμε λοιπόν στα πλαίσια αυτή τη βοήθεια να κάνουμε και στεναρές εκκλήσεις όπως πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να τονίσουμε κυρίως την ε, ελευθερία, την θρησκευτική. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι λίγο γενικόλογη διατύπωση. Στην Ιγυρία και όχι μόνο στην Ιγυρία είναι ιδιαίτερα θέμα θρησκευτικής ελευθερίας, ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης και δεν είναι μόνο αυτή η ομάδα που τόσο συχνά αναφέρθηκε που πρέπει να μας απασχολήσει, αλλά και η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι μόνο και μόνο από το ότι διαχωρίζουν την άποψή τους από την ε, δράση αυτή, ότι κατά δικά του δράση αυτή. Είναι μια χώρα με πολύ πληθυσμό, χρειάζονται λοιπόν πολύ περισσότερο από την κυβέρνηση στη χώρα της την ίδια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στάσνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταδικάζουμε όλοι τις ε, τρομοκρατικές ε, ε, επιθέσεις της Μποκοχάραμ κατά πολιτών, κυρίως δε χριστιανών. Είχαμε δύο επιθέσεις το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο με 250 νεκρούς και με μία ακόμα πιο έντονη κρίση ανάμεσα στον μουσουλμανικό βορρά και τον χριστιανικό νότο στην ε, χώρα χρειάζονται απεγνωσμένα και γρήγορα μεταρρυθμίσεις, διαρθρωτικές ε, αλλαγές. Ε, θα πρέπει να υπάρξει πολιτική, κοινωνική, οικονομική ανάπτυξη και αυτό σε όλες τις περιοχές γιατί είναι σημαντικός ο σταθεροποιητικός ρόλος της Νιγηρίας στην περιοχή αυτή. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι εθνοτικές και οι θρησκευτικές διαμάχες είναι βαθιά ριζωμένες ε, στην ε, ε, Νιγηρία και βεβαίως στοιχεία όπως η διαφθορά, η μη πρόσβαση σε πόσιμο νερό, η φτώχεια, η πανάπτυξη έχουν κάνει πιο έντονες αυτές τις διαδικασίες. Βεβαίως θα πρέπει να βοηθήσουμε και την κυβέρνηση της Νιγηρίας να εφαρμόσει κράτος δικαίου και ταυτοχρόνως να τιμωρήσει όσους έχουν ε, τελέσει τέτοιες, πράκτης, ε, τέτοιες πρακτικές. Ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε έτσι ώστε τέτοιου είδους ομάδες να εκριζωθούν, να μην υπάρχει πλέον αυτό το εθνοτικό ή θρησκευτικό μίσος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η Νιγηρία είναι η μόνη χώρα στον κόσμο ε, που έχει ίσο αριθμό μουσουλμάνων και ε, χριστιανών και μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προκλήσεις είναι να παραμείνει ενωμένη η χώρα και ταυτοχρόνως να καταπολεμήσει την τρομοκρατία. Έχουν γίνει πολλές επιθέσεις σε διοικητικά κτίρια, σε εκκλησίες κλπ. Ε, και ε, η επίθεση που έγινε στη διάρκεια της λειτουργίας των Χριστουγέννων σε μια εκκλησία είναι κάτι το αδιανόητο. Ο στόχος του κινήματος αυτού είναι να δημιουργήσει μίσος ανάμεσα στις διάφορες κοινότητες. Ο κύριος Μποχάρη, ε, ε, επικεφαλής των μουσουλμάνων, ε, έχει επικρίνει αυστηρότατα τις κινήσεις της κυβέρνησης του Προέδρου και κοινή τις ε, κοινότητες την μία κατά της άλλης ε, και μάλιστα τις ενθαρρύνει να ε, καταπολεμήσουν η μία την άλλη και συνολικά να καταπολεμήσουν τις δυτικές αρχές ξέρουμε, αρχές και αξίες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και διασυνδέσεις ανάμεσα στην Πόκο Χάρα και την Αλκάιντα. Γνωρίζομαι επίσης ότι υπάρχει σημαντικό ο όπλων προ την Νιγηρία από άλλες χώρες. Πρέπει να βοηθήσουμε πάση θυσία τη χώρα αυτή. Μπρόκ, το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, κύριε Επιτροπέ, πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό ή μάλλον να δούμε μαζί δύο πράγματα. Το ένα είναι κατά στην Ιγυρία, μια χώρα που είναι μέλος ΑΚΕ, όπου έχουμε καλές σχέσεις Κύριε Πίτροπε, ξέρετε, εσείς καλύτερα από μένα τη βοήθεια της δίνουμε, να λάβουμε επίση υπόψη μας, ότι η κυβέρνηση μιας πλούσιας χώρας που έχει τόσους φυσικούς πόρους είναι υπεύθυνη για να αξιοποιήσει τον πλούτο αυτό για καλύτερες κοινωνικές συνθήκες. Από την άλλη μεριά, η οργάνωση Μπόκο Χαράμ ε, χρησιμοποιεί μια γλώσσα που βλέπουμε και σε άλλες ε, μουσουλμανικές χώρες που χρησιμοποιείται από άλλες Ισλαμικές ομάδες, δηλαδή καταδιώκουν τους χριστιανούς. 75% των διώξεων για θρησκευτικούς λόγους αυτή τη στιγμή είναι κατά χριστιανών. Πρέπει λοιπόν να το διαπιστώσουμε. Ο Ισλαμικός κόσμος συνολικά, οι εκπρόσωποι του Ισλάμ, γιατί δεν υπάρχει μια κεντρική εξουσία, έχουν την υποχρέωση να διαφοροποιηθούν σαφώς από αυτές τις τάσεις. Είναι ο μόνος τρόπος. Το βλέπουμε στη Συρία, το βλέπουμε στην Αίγυπτο και βλέπουμε τι έγινε και στο Ιράκ. Και γι' αυτό είναι σημαντικό η εξωτερική υπηρεσία, η υπηρεσία εξωτερικών να ονομάσει έναν εκπρόσωπο για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που να ασχοληθεί με την ε, ε, καταδίωξη, με τις διώξεις των χριστιανών. Βεβαίως ε, υπάρχουν διώξεις για όλες ε, τις θρησκευτικέ ομάδες. Όλοι πρέπει να έχουν την ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης, αλλά εμείς ως Ευρωπαίοι πρέπει να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να διώκονται οι χριστιανοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα βλέπω τον κύριο Σουμάντσικη. Κυρίε και κύριοι, η Νιγηρία είναι μία ακόμη χώρα όπου το πολεμοχαρέ τμήμα του Ισλάμ θέλει δια τη βία να επιβάλλει τον Ισλαμικό νόμο. Το πρώτο θύμα αυτής της κατάστασης είναι οι χριστιανοί. Στο βόρεια, στη Βόρεια Νιγηρία γίνεται μια θρησκευτική κάθαρση με στόχο να εξολοθρευτούν οι χριστιανοί. Και μάλιστα η εφαρμογή της ΑΡΙΑ οδηγεί όχι μόνο μια εχθρότητα, αλλά και διακριτική μεταχείριση βάρος των χριστιανών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο σχολείο, στις ε, θέσεις εργασία και στην άσκηση της ε, θρησκευτικής λατρεία. Δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι απέναντι στα φαινόμενα αυτά. Θα πρέπει η διπλωματία μας να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να, κάνει να προστατεύσει την Νιγηρία από την αυξανόμενη θρησκευτική μυσαλλοδοξία. Θα πρέπει να εντείνουμε το διάλογο με την Νιγηρία και να ασκήσουμε ε, πολιτική πίεση ώστε κανένα στην Νιγηρία να μην πιστεύει ότι τα εγκλήματα κατά των εθνικών μειονοτήτων και ε, των θρησκευτικών κοινοτήτων θα παραμείνουν ατιμόρυτα. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε διαδικασία Catch the Eye και ο κύριος Μπρόνς. Η Νιγηρία <clears throat> παίρνει βοήθεια ακόμη 50 χρόνια μετά την ανεξαρτησία της. Δεν υπάρχει επαρκής οικονομική ανάπτυξη και οι περισσότεροι είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι τόσο φτωχή η Νιγηρία, μήπως επειδή δεν έχει πόρους. Όχι. Μα είναι η 8η μεγαλύτερη πετρέλαιο παραγωγός χώρα. Τι περίεργο. Επίσης υπάρχει ε, φίλια ένταση. Αυτό είναι εφημισμός για την ε, πίεση κατά των χριστιανών. Τι προκαλεί όλα αυτά τα προβλήματα, λόγω της φύσης του Ισλάμ, με την εθνότητα. Όχι, αυτά δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε φυσικά. Κάποιος Νιγηριανός που ήξερα είπα ότι είπε ότι έφταιγαν οι απεικιοκράτες που με ευθείε γραμμές δημιουργούσαν κράτη. Βέβαια αυτό σίγουρα συνέβαλε και συνέβαλε και στις αποσχεστικές τάσεις του 67. Αλλά εμείς οι Ευρωπαίοι δεν θα κάναμε το ίδιο λάθος. Δεν θα θέλαμε τα κράτη της Ευρώπης να έχουν διάφορους ασύμβατους πληθυσμού. Σίγουρα δεν θα το θέλαμε. Η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόσφατα ε, είχαμε πληροφορίες ε, για την ε, Νιγηρία σχετικά με μεγάλη βία. Μας απασχολεί περισσότερο η αύξηση ε, του, χριστιανικού, συγγνώμη, του θρησκευτικού φανατισμού μέσα από επιθέσεις κυρίως κατά των χριστιανών. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να αποφύγουμε την επιδείνωση της κατάστασης αυτής γιατί οι επιπτώσεις ε, ε, μπορεί να είναι καταστροφικές. 160 εκατομμύρια πληθυσμού έχει η χώρα αυτή. 50% του πληθυσμού είναι χριστιανοί και το άλλο 50% είναι μουσουλμάνοι. Η ε, ανάμεσα στις δύο αυτές ε, κοινότητες εντείνεται από την φτώχεια. Ε, είναι πολύ μικρό το κατακεφαλήν εισόδημα των Νιγηριανών, έστω και αν η Νιγηρία είναι σημαντική πετρελοπαραγωγός χώρα. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει προτάσεις έτσι ώστε να προωθηθεί το ερηνευτικό κλίμα στην χώρα. Ευχαριστώ. Θέλει κανεί, κανείς άλλος ad hoc το λόγο μέσω της διαδικασίας αυτής. Όχι. Οπότε παρακαλώ τον κύριο Επίτροπο. Αξιότιμα μέλη, πιστεύω ότι σήμερα για μία ακόμα φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε την ισχυρή του στήριξη προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαρκώς εμπλέκεται και περισσότερο στον εκδημοκρατισμό και την βελτίωση της κατάστασης στην Νιγηρία. Είναι γεγονός ότι βρίσκεται σε κρίσιμη ιστορική καμπή η χώρα αυτή αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα αλλά ταυτοχρόνως ανοίγονται μπροστά της και πολλές ευκαιρίες. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της Νιγηρίας. Αυτή τη στιγμή στηρίζουμε ε, την ε, ε, Νιγηρία με ένα ειδικό πρόγραμμα 200 εκατομμυρίων ε, ευρώ. Επίσης προσπαθούμε να βοηθήσουμε ιδιαίτερο στην περιοχή του Δέλτα ε, του Νίγηρα γιατί εκεί οι προκλήσεις οι αναπτυξιακές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Βεβαίως πρέπει να στηρίξουμε και την εκπαίδευση γιατί η Νιγηρία έχει έναν από τους πιο αρνητικούς δείκτες εκπαίδευσης 75 74% των παιδιών εγκαταλείπουν το σύστημα εκπαίδευσης. Είναι γεγονός επίσης ότι ε, η ε, Μπόκο εμποδίζει την νεολαία της ε, Νιγηρίας να εκπαιδευτεί, να βγει από την φτώχεια. Αυτό σημαίνει ότι δεσμευόμαστε απέναντι στην Νιγηρία και πρέπει να το κάνουμε με εντατικό ρυθμό. γίνεται συχνά λόγος στο διάλογο που έχουμε με την Ιγυρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, γίνεται λέω συχνά λόγος για την ελευθερία συνείδησης ε, και την ε, ελευθερία της θρησκείας. Αυτός ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ενδυναμωθεί στο μέλλον. Έχει δεσμευτεί η ίδια η ύπατη εκπρόσωπος και μάλιστα έχει και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες ε, τις οποίες ε, ε, ανέφερε και την προηγούμενη εβδομάδα στο, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στην Δανία. Έχουμε ξεκινήσει πλέον να δουλεύουμε την δέσμη μέτρων αντιμετώπισης της ε, τρομοκρατίας ε, έτσι ώστε να προσθεθεί αυτή η προσπάθεια στις διμερείς προσπάθειες που κάνουν ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να σταματήσει η έλλειψη απασχόλησης και η περιθωριοποίηση της κοινωνίας. Θέλουμε να εγκαθιδρυθεί ένα κράτος δικαίου θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη στρατηγική ε, κατά της τρομοκρατίας με ταυτόχρονο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, όσον αφορά τώρα τη δολοφονία των δύο Ευρωπαίων ε, ομήρων θα επαναλάβω για μία ακόμα φορά ότι εκφράζουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων για την τραγική τους απώλεια. Αυτές είναι εγκληματικές πράξεις. Ε, η ε, σύλληψη, ε, η εγμαλώτηση ομήρων είναι σίγουρα εγκληματική πράξη την οποία καταδικάζουμε. Τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι τα έσοδα από, την, από τις εξαγωγές πετρελαίου. Έχει γίνει ήδη πρόταση για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις προσόδους από, τις, από τους φυσικούς πόρους της χώρας και βεβαίως θα στηριχθούν τα μέτρα αυτά γιατί καταλαβαίνουμε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος της ε, ένδυας σημαίνει ότι θα πρέπει όλες οι πετρελαϊκές ε, ε, εταιρείες με διαφάνεια να προωθούν τα οικονομικά τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Έχουν υποβληθεί 7 προτάσεις ψηφίσματος για το θέμα αυτό από τις πολιτικές ομάδες. Κλείνει η συζήτηση για την Ιγυρία. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, χωρίς διακοπή, την κατάσταση στη Λευκορωσία. Οπότε, παρακαλώ τον Επίτροπο Πίμπαλξ ως εκπρόσωπο της ΙΑΠ, κυρία Σάστον. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Μεγάλη μου χαρά ε, να συζητήσω σήμερα την κατάσταση στην Λευκορωσία από πλευρά τη υπάτη εκπροσώπου κυρία Άστον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί όλο και περισσότερο για τη συνεχιζόμενη